start. I'm ready. Cari colleghi, Αγαπητοί συνάδελφοι, με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε την Βία Κέλ που είναι συνάδελφος ε, βουλευτής στο Ιρακινό Κοινοβούλιο. Κανείς